εξέταση του επόμενου σημείου της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος έχει λάβει από την ε, ομάδα του ΕΛΚ ένα αίτημα ορισμού υποψηφιότητα σε μια αντιπροσωπεία. Ο διορισμός αυτός θα υπάρξει στα πρακτικά και αν δεν γίνουν και δεν υποβληθούν παρατηρήσεις μέχρι τη στιγμή της έγκρισης των πρακτικών, ο διορισμός θα θεωρηθεί ως κάτι που έχει γίνει αποδεκτό. Πρόκειται για τον κύριο Ντάριο Ροζάτη που προτείνεται να αποτελέσει μέλος της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euron. Αυτό καταρχάς. Έρχομαι τώρα